για την εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων και θα ζητήσω από τον Επίτροπο κ. Μουέντας να λάβει και πάλι το λόγο εξ ονομάς Κομισιόν. Κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη. Ο Επίτροπος Κανιέται <clears throat> λυπάται που δεν μπορεί να έρθει εδώ. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση για τις μεθόδους υπολογισμού και τις ανάγκες αναφορών σε σχέση με το άρθρο 7α της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων μπορεί να περατωθεί αυτή η διαδικασία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να μπορέσουν να αρχίσουν να εφαρμόσουν αυτό το στοιχείο του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν τα μέτρα μετριασμού των αποτελεσμάτων τη κλιματική αλλαγή για να επιτευχθεί ο στόχο 6% μείωση των αερίων θερμοκηπίου από τα καύσιμα το 2020. Το Συμβούλιο επέτυχε την ειδική πλειοψηφία σε σχέση με την πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν τον Οκτώβριο. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η πρόταση και θεωρούν ότι δεν θα μπορέσει να μειώσει τη χρήση μη συμβατικών μορφών ε, καυσίμων όπως από τις ασφαλτούχες άμμου να έρθουν, άμμους να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η, σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος του άρθρου 7α της οδηγίας είναι να μειωθεί η χρήση του περιεχομένου άνθρακα στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για μεταφορές. Ο στόχος δεν είναι να αποθαρρύνουμε τη χρήση οποιοδήποτε είδους καυσίμου, αλλά να εξασφανίσει ότι θα υπάρξουν τα απαραίτητα μετριαστικά μέτρα ώστε να επιτύχουμε το στόχο 6% μείωσης της εκπομπής αερίων από καύσιμο από το 2020. Η Κομισιόν επεπισμένη ότι η οδηγία για τα, την ποιότητα του καυσί, των καυσίων μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη σε αυτή την πρόταση. Η νέα πρόταση της Κομισιόν που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο έχει ένα χαρακτήρα εξισορροπημένης συμβαστικής λύσης γιατί επιτυχάνει τους στόχους της βασικής πράξης αλλά λαμβάνει υπόψη και τις ανησυχίες των κυρίων εμπλεκομένων με σωστό τρόπο. Η Κομισιόν όμως είναι έτοιμη να, εξετάσει, να επανεξετάσει την εμπειρία για την εφαρμογή του άρθρου 7α ως τμήμα του προγράμματος της καλής ρύθμισης επέκεινα και του 2020. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι επιλογές για να μπορέσει να μειωθεί το επίπεδο των εκπομπών από καύσιμα για μεταφορές και να επιγραμμιστεί με τον στόχο μιας μείωσης τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030. Όλοι οι εμπλεκόμενοι και εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσκληθούν να αναφέρουν τις απόψεις τους μέσα σε μια συνδιάσκεψη που θα διοργανωθεί το 2015. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για τρία λεπτά κύριε Γκύρκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις κλιματολογικές αλλαγές και ένα τμήμα των προσπαθειών αυτών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Είμαστε σε αυτό πρωτοπόροι διεθνώς στον αγώνα αυτών κατά των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, τους στόχους αυτούς, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα της βιομηχανίας, να μειώσουμε τα γραφειοκρατικά άχθη, να διασφαλίσουμε μεν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και να διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα της υπήρου μας. Η Κομισιόν θέλησε να εξισορροπήσει τα δύο αυτά στοιχεία με την πρότασή της και θα ήθελα να προσέξετε και εσείς συνάδελφοι το γεγονός ότι καταψηφίζοντας τη συμβιβαστική αυτή πρόταση θα τεθεί σε κίνδυνο η δουλειά πέντε ετών γιατί είναι αποτέλεσμα μακράς διαπραγμάτευσης και μπορούμε με το συμβιβασμό αυτό επιτέλους να αρχίσουμε να καταπολεμούμε τις εκπομπές διοξιδίου τα επίπεδα των εκπομπών πρέπει να αναφέρονται. Σωστό αυτό. Αλλά η πρακτική του εφαρμογή δεν μου φαίνεται ρεαλιστική γιατί είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η αυθεντικότητα των στοιχείων που θα χορηγούν οι βιομηχανίες και επίσης να επιτευχθεί η πιστοποίηση γιατί θα σήμαινε αυτό δυσανάλογο γραφειοκρατικό άχθος και θα επηρέαζε, θα στρέβλωνε και τον ανταγωνισμό. Όσοι δεν θέλουν να εισάγουν καύσιμα από τον Καναδά, ας πούμε, θα τιμωρούνται. Κάτε με, ο μέσος δείκτης είναι πολύ καλό εργαλείο για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέσων. Γι' αυτό προτείνω να δεχτούμε τη συμβιβαστική πρόταση της Κομισιόν. Αν την απορρίψουμε τότε θα καταστρέψουμε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του 6%. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκρότ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την ποιότητα των καυσίμων και μας ελέγχεται ότι είμαστε μη ρεαλιστές. Από το 2011 μέχρι το 2040 θέλουμε να μειώσουμε κατά 40% θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του περιβάλλοντος. Όχι. Εγώ θέλω να σας προειδοποιήσω. Αν τα πράγματα προχωρήσουν και στο μέλλον με τον τρόπο αυτό, ώστε οι ρυθμίσει του πακέτου ενέργειας και κλίματος αλλάζουν, αντί να βελτιωθούν, τότε μπορούμε να πάμε σπίτι μας, γιατί ουσιαστικά θα μας κοροϊδεύουν πια στο μέλλον και θα γινόμαστε περίγυλος, περίγυλος της διεθνής διαπραγματεύσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια λύση να δώσει μια δήλωση η Κομισιόν και χαίρομαι που είσαστε παρόντες, αλλά περίμενα να έρθει κάποιος άλλος ή μάλλον δύο άλλοι να ερχόντουσαν εδώ. Πάλι καλά που είσαστε εσείς και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να έρθει εδώ με μια σαφή δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο θα, η, θα φερθεί στην συνδιάσκεψη για το ε, για τη διάσκεψη για το κλίμα. Δεν μπορούμε να λέμε μία μέρα το α και την άλλη μέρα το άλλο γιατί αυτό που θα κάνουμε θα είναι το υπόδειγμα για όλους τους διεθνείς εταίρους μας. Εμείς θα πρέπει να θεσπίσουμε λοιπόν τα πρότυπα και πρέπει να αγωνιστούμε για να επιβάλλουμε τη θέλη μας και τελικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι οριακές τιμές θα προχωρήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε μειώσεις και εκτός σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Κρότε. Η κυρία Γκίρλιν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Γκρότε λέει μόνο όχι μπορούμε να πούμε. Μα αυτή η απόφαση αντιμετωπίζεται μέσα από τη διαδικασία ρύθμισης με έλεγχο. Γιατί είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας οποιαδήποτε αντίρρηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Δεν αρκεί να πούμε ναι ή όχι. Πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση για ένα από τρει λόγου. Και αυτοί που προτείνουν την αντίρρηση έχουν προτείνει τον ε, αποχρόντα λόγο υποαριθμό 3. Αλλά αυτό είναι ασύμβατο με το περιεχόμενο τη δράση. Είναι σαν να λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει σωστή αναφορά του όγκου και τη ποιότητα και των χαρακτηριστικών των καυσίμων. Βέβαια, δεν προχωράει αυτή η πρόταση τόσο πολύ όσο θα θέλανε ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά τα στοιχεία, η τεκμηρίωση για το σημείο 3 δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά για την πρόταση τη Κομισιόν. Η πρόταση αυτή ζητάει από τι μεγάλε εταιρείε να αναφέρουν από πού εισάγουν αργό πετρέλαιο. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στον καταναλωτή και αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στην ε, κοινή γνώμη. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει πιο εύκολη ενημέρωση των στοιχείων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο μέλλον. Και με την οδηγία αυτή η οποία δεν περιλαμβάνεται στους ε, στόχους του, της Κομισιόν επέκεινα του 2020 η έγκριση αυτής της αντίρρησης θα υποσκάψει μονάχα την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη θεσμική καθυστέρηση για ένα θέμα το οποίο η ρύθμισή του θα εκπνεύσει σε έξι χρόνια. Αυτό δεν θα είναι θετικό. Η καλύτερη λοιπόν συμβαστική λύση που θέλει ο κύριος Χρότε, η καλύτερη συμβαστική λύση λοιπόν είναι το Κοινοβούλιο να προχωρήσει με την πρόταση Κομισιόν και να τη δεχτούμε ως ένα θετικό βήμα και να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε κάπου τα επόμενα χρόνια και να μην το αφήσουμε αυτό το θέμα εκρεμές σε διαθεσμικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Χερμπράντι για δύο λεπτά. Thank you, Madam Chair. It was this week... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το Σαββατοκύριακο επέστρεψα από τη Λίμα, όπου έλαβε χώρα η διάσκεψη κορυφής για το κλίμα. Ε, ε, και θα πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα με την αποφασιστικότητα ε, με την οποία αντιμετωπίζονται οι κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα τη διάσκεψη αποδεικνύουν ότι ο αγώνας μπροστά θα είναι δύσκολος. Ο κόσμος θα εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα αύριο και ακόμη περισσότερο μεθαύριο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα οικονομία και μετά να περάσουμε στην ε, οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Με συγχωρείτε, λέει ο μιλητής. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα, στις διάφορες ε, ε, ζωοτροφές ε, και με συγγνώμη, σε διάφορα προϊόντα καυσίμων, ας πούμε τα πολύ ε, μο, ε, χειρότερα σε ποιότητα νιγηριανό πετρέλαιο ε, τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης με άλλα πολύ καλύτερα διελισμένα ε, πετρέλαια από άλλους προμηθευτές. Ε, είμαι πολύ απογοητευμένος από τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν σήμερα, γιατί εγώ ανέμενα ένα, μια πολύ πιο στεναρή δέσμευση στους στόχους της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, αφού είδα την πρόταση του 2011, πώς μπορείτε τώρα να υπερασπίζεστε μια τελείως αντίθετη πρόταση αφού απέρριψε την πρώτη σας πρόταση το Συμβούλιο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε να τα υποστηρίζετε και τα δύο, αφού είναι απόλυτα σαφές ότι πρέπει να κινητοποιηθούν, να αναζωπηρωθούν οι επενδύσεις και αυτό μπορεί να γίνει μόνο προς τη σωστή κατεύθυνση, αν τις ενθαρρύνουμε να γίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και αντίθετα τις αποθαρρύνουμε από το να, να πάρουν τη λάθος κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γερμπράντη. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Λόπες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν η πρόταση του Συμβουλίου να, να συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις ελευθέρω εμπορίου με τον Καναδά γιατί το κείμενο αυτό συμπίπτει απόλυτα με αυτά τα οποία ήθελε το πετρελαϊκό λόμπι να ανοίξουμε τελείως την αγορά στα καύσιμα από τους, τις ασφαλτούχους άμμους του Καναδά. Αυτό όμως το καύσιμο οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το λέει και η ίδια η, η έκταση της Κομισιόν είναι πραγματικά τρομερό το ότι δεν θέλουν καν να, να αντιμετωπίσουν το πετρέλαιο αυτό το οποίο είναι τόσο αρνητικό. Η συμφωνία που θέλει να κάνει λοιπόν η Κομισιόν και το Συμβούλιο με τον Καναδά και το, τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά αυτό το κάνουν σε βάρος των προστασιών που υπάρχουν στο περιβάλλον, για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται όλο και μεγαλύτερη η αντίφαση στις πολιτικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν εφαρμοστούν σωστά αυτέ πολιτική, η συσσόρευση κέρδους είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ακυρώνει την αποτελεσματικότητα. Όλο και περισσότερο μπαίνουμε σε μια παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας η οποία είναι ε, αφόρητη σε επίπεδο βιωσιμότητας για το περιβάλλον και τους καταναλωτές γίνεται ουσιαστικά μια διαδικασία η οποία οδηγεί και στην καταλήστευση γεών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια βιώσιμη εναλλακτική λύση και όχι αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκχάουτ για τέσσερα και μισά λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούμε από παντού ότι η αντίρρηση δεν είναι για την οδηγία ποιότητα των καυσίμων. Εμείς είμαστε υπέρ της οδηγίας. Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματικό όπλο, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, θεωρητικά. Γιατί με την πρότασή της αυτή η Κομισιόν ηθελημένα αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητά της. Και αυτό το λέω και στον συνάδελφο Γκέλιν που είπε ότι μόνο για νομικούς λόγους μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση. Αλλά διαβάστε την αξιολόγηση και θα δείτε ότι η θελημένα η Κομισιόν αφαιρεί ένα από τα όπλα για την επίτευξη του στόχου του 6%. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ ζωοτροφών που είναι ένας από τους τρόπους μείωσης. Άρα αφαιρεί την αποτελεσματικότητα ενός από τα δυνατά μέσα. Γι' αυτό είμαστε κατά. Επίσης, άμα διαβάσετε την μελέτη αντικτύπου, θα δείτε ότι ενώ αύριο η Κομισιόν θα μας κάνει προτάσεις για καλύτερη αποτελεσματικότητα, παρόλα αυτά η πρόταση του 11 είναι η πιο αποτελεσματική. Είχε γίνει και τότε μελέτη αντικτύπου. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν δεν ακολουθεί την ίδια της την αξιολόγηση την ίδια της την πρόταση του 11 έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα από τότε όχι άμα δείτε τη μελέτη αντικτύπου θα δείτε ότι όλες οι τιμές είναι οι ίδιες όπως το 11 άρα μπορούμε να μαντέψουμε τι συνέβη και καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με τον συνάδελφο Ματίας Χόλτερ είναι αποτέλεσμα τη καναδικής πίεσης τα καναδικά λόμπι θα έχετε λάβει κι εσείς μάλλον ηλεκτρονικά μηνύματά του να υποστηρίξουμε την πρόταση γιατί, γιατί τώρα δεν διαφοροποιούμε αυτά που πρέπει να διαφοροποιηθούν. Άρα εδώ πέρα απλώς υποστηρίζουμε με την πρόταση αυτή το καναδικό λόμπι. Και μάλλον θα μας ακούν οι Καναδοί τώρα. Αυτό δεν το λέω κατά του κράτους του Καναδά. Εμείς θέλουμε διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων τύπων καυσίμων. Αν μπορούν να μας δείξουν οι Καναδοί, να μας αποδείξουν ότι μπορούν να παραγάγουν με καθαρό τρόπο καύσιμα, θα το αναγνωρίσουμε. Θέλουμε λοιπόν την διαφοροποίηση. Τα πιο μολυντικά καύσιμα να τα ξέρουμε ποια είναι και τα λιγότερο επίσης. Και δεν το λέει αυτό η πρόταση η τωρινή. Άρα καταπολεμά τους στόχου της η οδηγία. Ήλπιζα να είχε καταλάβει η Κομισιόν ότι η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων είναι κάτι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, τι μας είπε, απλώς θα αναθεωρήσουμε, θα οργανώσουμε ένα συνέδριο, αυτά. Όχι, εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω. Πώς θα διασφαλίσει η Κομισιόν ότι μέχρι το 20 θα υπάρξει πρόταση που να λαμβάνει υπόψη της τη διαφοροποίηση των τύπων καυσίμων ώστε να επιβραβεύονται τα μη μολυντικά και να τιμωρούνται τα μολυντικά. Είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚΑ αν την απορρίψουμε την πρόταση θα χαραμίσουμε πέντε χρόνια προσπαθειών. Όχι, άμα την εγκρίνουμε θα χαραμίσουμε την προσπάθεια. Είναι μια κενή πρόταση. Αν σας ενδιαφέρει όντως η σωστή μεθοδολογία τότε πρέπει να πολεμήσετε κι εσείς υπέρ της προηγούμενης πρότασης του 11 που διαφοροποιούσε τα καύσιμα. Υπάρχουν κι άλλα λόμπι βέβαια όπως των βιοκαυσίμων αλλά δεν λέω ότι αυτή είναι καλή και η Καναδή κακή λέω ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η σωστότερη πρόταση. Επομένως αυτή είναι η αντίρρησή μας και δυστυχώς κύριε Επίτροπε δεν μας επιτρέπετε, δεν μας αφήνετε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να καταψηφίσουμε δυστυχώς αυτή την πρόταση με πόνο ψυχής. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παιδικίνη για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ εγκρίνω τα όλα όσα είπε ο συνάδελφο Εκχαούτ. Να προσθέσω μόνο κάποια τεχνικά στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι όλε. Δεν, δεν είναι όλα τα καύσιμα καταστρεφτικά για τον άνθρωπο και για το και περιβάλλον, αλλά ακόμα ε, πιο καταστρεπτικά είναι η ε, ασφαλτούχες αλλά και το αέριο από σχιστόλιθο. Έχουν, υπάρξει, έχουν ληφθεί δείγματα όπου είναι 6.000 φορές ψηλότερη περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια η <coughs> περιεκτικότητα ε, σε σωματίδια, όπως είπα, στις περιοχές όπου έχουν χρησιμοποιηθεί αυτού του είδους τα καύσιμα και στις κλινικές βλέπουμε ε, αύξηση λευκαιμίας, ε, ειδικά από τη στιγμή που προχωρούσαμε πιο κοντά στις περιοχές που είναι μολυσμένες από αυτού του είδους τα καύσιμα. Δεν λαμβάνει η Κομισιόν υπόψη αυτό, αυτές τις μετρήσεις που έχουν γίνει για τις ασφαλτούχες και για το αέριο από σχιστόλιθο. Πώς ε, αντέχετε ακόμα αυτή την Κομισιόν που κάνει τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ τους συμπολίτε μου. Ευχαριστώ κύριος Γιάουκ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο αγώνας κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας και της μείωση των αερίων θερμοκηπίου είναι μια από τι μεγαλύτερε συζητήσει σε επίπεδο οικολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπω το κατεχνεί και η διάσκεψη τη Λίμα που τελείωσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι απαραίτητο να ξεπεράσουμε το στάδιο των ευχολογίων και των καλών προθέσεων. Όμω αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Αν ήταν πιο λιγότερο σοβαρό το θέμα, θα έλεγα ότι το θέμα αυτό γίνεται απλό ως μια μεξικανική λύση, μια περουβιανή λύση. Στη Λίμα με την ε, υπόθεση ότι θα υπάρξει μια συμφωνία το 2015 στο Παρίσι, μιλάμε για το φύλλο των αγγέλων. Ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα που να εξασφαλίσουμε ένα πιο ευέλικτο πρωτόκολλο για τι αναπτυσσόμενες χώρε. Η οδηγία της Κομισιόν που συζητούμε σήμερα είναι από τα κομμάτια της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια. Η Κομισιόν προτείνει πέντε κυρίους άξονες για τους περιορισμούς που θα παραγωγιστούν στους παραγωγούς καυσίμου για να μειωθεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Βασίζεται σε πολύ τεχνικά στοιχεία υπολογισμού. Και αυτό είναι ο υπολογισμό της Κομισιόν που διαφυσβητείται από τους κύριους Χερβράνδη και Εικ Χάουτ. Οι δύο πλευρές εδώ έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο. Και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν υπερβολικά μαθηματικές και νομικές θεωρήσεις για να κρύψουν τις παραταξιακές τους απόψεις, οι οποίες δίνουν, έχουν μεγαλύτερη σημασία από την οικολογική λύση. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει η υπολογισμοί αυτή να μην είναι αυτοί που θέλει η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής. Ο Καναδός Υπουργό Φυσικών Πόρων έχει ήδη στραφεί εναντίον μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία θέλει να διατηρήσει τους παραδοσιακούς πετρελαϊκούς πόρους για την αντίληση αυτή που έχει διατυπωθεί βάσει του άρθρου 106 του κανονισμού ψάχνουν ένα πρόσχημα για να μπορέσουν να <clears throat> ε, ξεχωριστούν από την πτέρυγα αυτή που έχει υποστηρίξει το Jean-Claude Juncker και έχει χάσει την αξιοπιστία της. Επομένως δεν μπορεί να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Η πολιτική μας θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες γενικού συμφέροντος και όχι τον μερκαντιλισμό. Ο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν πρόκειται για μια αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τα καύσιμα. Θα πρέπει αντίθετα να βελτιώσουμε αυτή την οδηγία και εγώ συμφωνώ με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν. Τι σας οδήγησε να κάνετε αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης. Έχετε κάνει αναλύσεις που καταδεικνύουν ότι οι ασφαλτούχες άμοι και τα καύσιμα που παράγονται από εκεί επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το κλίμα από άλλες μορφές ενέργειας. Τι σας έχει κάνει να αλλάξετε λοιπόν την αντιμετώπιση σας ή μήπως άλλαξε απλώς η πολιτική σας. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει δεκτό γιατί δεν υπάρχει καν καμία επιχειρηματολογία γιατί πρέπει να δεχτούμε αυτό. Ξέρουμε ότι τα καύσιμα για τις μεταφορές έχουν μεγάλο ρόλο στην εκπομπή ε, αερίων θερμοκηπίου και είδαμε στη δεκαετία του 1990 ότι ήρθαν και πιο βρώμικα καύσιμα στην αγορά λόγω ακριβώς αυτής της οδηγίας και λόγω των νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την ε, ε, χρήση πετρελαίου από ασφαλτού για σάμους και αερίου από τους. Η οδηγία αυτή κανονικά θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαφοροποίηση αυτών των ε, πηγών ενέργειας. Δεν πρέπει λοιπόν να γονατίσουμε μπροστά στα πετρελαϊκά όπλα, ο, πετρελαϊκά λόμπι. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο. Γιατί και άλλοι θα ακολουθήσουν κάτι τέτοιο. Στο τέλο δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε πολιτικό επίπεδο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Απλώ θα υποκύπτουμε στα πελατειακά συμφέροντα. Αυτό είναι ανάξιο του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλό το κόστο για του συμμετέχοντε στην αγορά. Στην εποχή του ίντερνετ δεν είναι καθόλου δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις στη τιμή των καυσίμων. Θα πρέπει λοιπόν να απορρίψουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί η πολιτική μας. Ο κύριος Τόρβαλς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτή η πρόταση είναι ταυτόσιμη με το έγγραφο που έχουμε ειδηθεί και στην τρίτη σειρά περιλαμβάνεται μια υπόσχεση και την παραθέτω μια πολιτική για το κλίμα ε, που θα είναι πιο μακροπρόθεσμη. Όμως ας δούμε μια σύντομη ματιά, με μια σύντομη ματιά την ιστορία. Πριν από τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την ε, διάσκεψη της Κοπενχάγης ε, για το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια. Η οδηγία περί ποιότητας των καυσίμων είναι η μόνη νομοθεσία από αυτό το πακέτο που δεν έχει εφαρμοστεί. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το 2020 είναι σχεδόν εδώ και ότι πλησιάζουμε στη διάσκεψη του Παρισιού που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο, χρειάζεται ισχυρή εφαρμογή αυτής της οδηγίας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς ε, την ε, κοινωνία χαμηλού, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα που θέλουμε. Για να έχει νόημα κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ακρίβεια και στην εφικτότητα. Σωστή καταμέτρηση λοιπόν των εκπομπών είναι πολύ θεμελιώδης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι πίσω και οι σχετικές επενδύσεις έχουν παγώσει οι αναπτυξιακές πολιτικές ε, και η ανάπτυξη σε βιομηχανίες που καταναλώνουν και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα δεν θα είναι η λύση. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ρίντ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι ευτυχή που λέω για μια φορά ο απλό άνθρωπος ωφελείται από τις διεθνείς εξελίξει. Οι τιμέ του πετρελαίου και του φυσικού αερίου πέφτουν. Και αυτό γιατί χώρε, όπως είπα και ο Καναδάς ανοίγουν νέου ε, πόρους και μειώνουν το κόστος της ενέργειας. Ένα αποτέλεσμα είναι ότι εξαρτώμεθα λιγότερο από ασταθείς χώρες και εχθρικά καθεστώτα. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ότι το κόστος του καυσίμου μειώνεται που, για τον κόσμο που πιέζεται από τη λιτότητα. Καλά νέα για τον καινούριο χρόνο, αλλά όχι βέβαια αν είσαι πράσινος που θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν για να τορπιλήσουν αυτές τις εξελίξεις. Η Κομισιόν δεν προτείνει καμιά συμφωνία για τη θέσπιση στόχων για να μειωθεί ή και για να ψηφιστεί ο κόσμος ε, που έχει ξεζουμιστεί. Είναι δύσκολο ε, γιατί δημιουργήθηκε ένα νόμισμα με ένα σωρό δομικά μειονεκτήματα και μειώθηκε, μειώθηκαν οι συνθήκε διαβίωση εκατομμυρίων. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγέ. Τα πρόσφατα χρόνια το κλίμα αρνείται να αντιστοιχήσει, να αντιστοιχηθεί μάλλον στις αποκαλυπτικές ε, προβλέψεις και προφητείες. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σβάνη για ένα λεπτό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που σε αυτή τη μακρά συζήτηση που διερκεί πάνω από πέντε χρόνια, που διαρκεί μάλλον ότι και πέντε χρόνια, ισχυρίζονται ότι αυτή η πρόταση της ε, Κομισιόν έχουμε πολλές φορές σκοντάψει. Η πραγματική λύση δεν είναι απαραίτητο η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η πραγματική λύση είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει, εξορίσεται από την ε, γη, αλλά παράγεται πάνω από την επιφάνεια της γης. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές οι οποίες δεν θα προκαλέσουν πια αυτές τις αντιφάσεις και τις αντιρρήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κυρία Μπίρντερ, είναι πολύ απογοητευτικό που η Κομισιόν αισθάνθηκε πίεση να προτείνει μια αδύναμη απάντηση όσον αφορά τι ασφαλτούχε άμμουσε στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία. Αγνοούνται διάφορε συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα είδη ε, καυσίμων. Η Κομισιόν επίση έχει αποτύχει να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα τη δική τη ε, εξολόγηση κινδύνου. σε αποτέλεσμα, οι ασφαλτούχες άμμος ε, θεωρείται ε, το ίδιο όπως τα συμβατικά καύσιμα και οι εταιρείε δεν θα μπορούν να αναφέρουν ούτε καν εθελοντικά τις πραγματικές εκπομπές των καυσίμων τους. Ε, αντί να επενδύει σε καθαρότερα καύσιμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει τι πόρτες της για την τις ε, πολύ βρώμικες ασφαλτούχες άμμους αλλά και το πετρέλαιο. Επιτρέπει την εισαγωγή ασφαλτούχου άμμου από τον Καναδά. Παρακαλούμε αγαπητή Κομισιόν να αναπτύξετε νέα μέτρα ώστε να παραταθεί η οδηγία ποιότητας των καυσίμων πέρα από το 2020 λαμβάνοντας υπόψη πόσο πολύ ρηπαίνει η ασφαλτούχο είχε άμμος αλλά και το ακάθαρτο πετρέλαιο. Αν πραγματικά νοιαζόμαστε για τι κλιματικέ αλλαγέ και για την προστασία του περιβάλλοντο, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί για τη μείωση των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών και αυτό μπορούμε μόνο να το καταφέρουμε αν ξέρουμε τι καίμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Η επομένη είναι η κυρία Λαουρίστεν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να προσέξει και κάτι άλλο σε σχέση με αυτή την οδηγία. Γιατί το θέμα εδώ δεν είναι μόνο το τι γίνεται στον Καναδά, αλλά και το τι γίνεται και με τους παραγούς καυσίμων στην Ευρώπη, οι οποίοι πασχίζουν να έχουν καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό ισχύει και στην Εστονία. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες να μπορέσουμε να έχουμε περιβαλλοντικό το συμπίν, φύλλο περιβαλλοντικό τέλο πάντων καύσιμο και πετρέλαιο συγκεκριμένα. Οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς έτσι θα βρούμε και τις πασχόλησεις για χιλιάδες Έτσι ε, Και έτσι έχουμε λοιπόν και τη μειονότητα. Οπότε και αν αποδορυφθεί αυτή η οδηγία για τη χώρα μας θα σημαίνει ανεργία. Θα διπλασιαστεί η ανεργία και μιλάμε για έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Κοινωνική αναταραχή θα έχουμε. Γιατί μιλάμε για μια περιοχή κοντά στην Μερθόριο με τη Ρωσία, που πηγαίνει το όλο και πιο επιθετική. Άρα και αυτό λάβετε υπόψη. Αλλά είναι και περιβαλλοντικό το πρόβλημα είναι και κοινωνικό και στρατιωτικό. so much, young might... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι νέος και αφελήσα και εξακολουθώ να πιστεύω σε ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό με πληγώνει όταν βλέπω πως ε, μετά από τέσσερα χρόνια τα πράγματα χειροτερεύουν. Οι προτάσεις που έχουμε τώρα ε, ε, επιτάπητος είναι χειρότερες από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια η ΔΕ Κομισιόν αφαιρεί τα κίνητρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί πρέπει να πιστέψουμε πως υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν απαγορεύουμε κανένα καύσιμο. Τι λέμε, χρειαζόμαστε διαφορετικούς κανονισμούς για να δώσουμε κάνα κίνητρο να βελτιωθεί η κατάσταση. Και φοβάμαι πως αυτό που βλέπουμε είναι σημάδι της νέας Κομισιόν και θα μας πούνε αύριο πως πάρα πολλά θέματα του περιβάλλοντος θα αποσυρθούν. Ελπίζω να κάνω λάθος ε, και να αποδειχθεί πως έχω λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. πρόταση της Κομισιόν για την ποιότητα των καυσίμων παρουσιάζει πολλές ελλείψεις. Δεν επιτρέπει διαφοροποίηση ανάμεσα στα θέματα των διαφορετικών πρώτων υλών και ούτε καν η ανακοίνωση για την πραγματική, τις πραγματικές Με βάση τις μεθόδου που έχουμε κάνει, τα, τα καύσιμα εκτιμώνται χαμηλότερα από την πραγματική τους αξία και εκ τούτου ευνοείται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό το φως αυτών των στοιχείων βλέπουμε ότι η ένσταση που έχει υποβληθεί στην πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να θεωρηθεί θεμητή. Αλλά πιστεύω πως για την εξολόγηση της της Κομισιόν δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το γενικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται, δηλαδή το θέμα της, ε, ε, ε, ε ασφάλειας ε, ε, του ανεφοδιασμού της Ένωσης. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να ευνοήσει την, ε, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που θα βελτώνουν την αποδοτικότητα των καυσίμων. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των ομάδων, η κυρία Μάισνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. πρέπει να μειωθεί κατά 6% η ένταση των καυσίμων στον κύκλο ζωής τους ε, όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δυστυχώς αντί να γινόμαστε πιο φιλόδοξοι, γινόμαστε λιγότερο φιλόδοξοι. Και εδώ πέρα βλέπετε πως η ένταση διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθεί και αυτό προτείνεται ως συμβιβασμό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το εξής για το τι μπορούμε να πούμε κατά σε αυτό το οποίο είπατε. Εντάξει, έχει μεγάλη σημασία και η εξάρτηση από εισαγωγές και το τι θα κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις σύνον Καναδά και εγώ θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε κάποια απάντηση γεγονός είναι πως ε, προφανώς ε, οι φιλόδοξοι στόχοι πλέον δεν ε, ισχύουν. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην διαδικασία του ΚΕΤΣΔΙΑΗ για λίγα λεπτά. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Φλασίκοβα. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως είναι σημαντικό να περιοριστούν πράγματι οι εκπομπές του διοξιδίου του ανθρακά και να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020 πράγματι Ε, αυτό δεν μας δείχνει κάποια προσπάθεια περισσότερης αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με ρεαλιστικούς στόχους. Εμείς θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο την επιδείνωση. Είμαι σίγουρη πως η Κομισιόν θα μπορούσε να συντάξει μια θέση την οποία θα στηρίξει το Κοινοβούλιο και να μην υποκύψει στην πίεση των λόμπι. απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν να κάνει μια καλύτερη έκθεση. Η Κομισιόν μπορεί να κάνει μια σαφή πρόταση σύμφωνα με αυτό που αποτελεί ή είναι μάλλον το κλειδί των προσπαθειών στην καταπολέμηση λοιπόν της κλιματικής αλλαγής φυσικά και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αλλά και η προστασία των καλαρωτών έχει ύψιστη σημασία. Όταν ε, συζητάμε για σοκολάτα μιλάμε για την υγεία του καταναλωτή. Εδώ μιλάμε για καύσιμα που ε, χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες της Ένωσης και ε, μας επηρεάζουν όλους. Φυσικά θα πρέπει να προχωρήσουμε με στόχο την πράσινη οικονομία, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, οικονομίες ε, των, των κρατών από τις οποίες κάνουμε εισαγωγές. Ευχαριστούμε επόμενη αγορήτρια κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ. Υπάρχει υποκρισία στην ε, συζήτηση αυτή. 94% του τομέα των μεταφορών εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα. Και η Κομισιόν μας λέει εδώ πέρα πως ε, το μέτρο αυτό δεν στέκει νομικά και δεν είναι κατάλληλο. Μα πρώτα απ' όλα επενδύουμε στην έρευνα και την τεχνολογία. Και όμως ασχολούμαστε και τσακωνόμαστε για κάτι το θετικό όπως αυτό το μέτρο. Γελία κατάσταση δηλαδή. Συγκεκριμένα το εκτιμώντας 44 της οδηγίας ε, πώς είναι δυνατόν να λέμε πως το να ενισχύουμε τα υφιστάμενα δεν είναι στόχος της οδηγίας που στόχο έχει να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τα καύσιμα. να συντονιστούμε λίγο. Και εγώ συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους των σοσιαλιστών και άλλους. Ευχαριστώ κυρία Καλάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε το τι θέλουμε εδώ να πετύχουμε. Τη μείωση δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η Εστονία έχει την ιδιαιτερότητα του να έχει ε, έναν τέτοιο κλάδο σχιστολιθικού αερίου ο οποίος ρηπαίνει, γι' αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα. Αν απορρίψουμε την πρόταση Κομισιόν κινδυνεύουν οι επενδύσεις που έχουν γίνει και θα οδηγηθούμε σε περισσότερη ρήπανση. Το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία επίσης πρέπει να το έχουμε κατά νου. Η απόρριψη της πρότασης θα οδηγήσει σε μετατόπιση της παραγωγής και των θέσεων εργασία από την Εστονία στη Ρωσία. Και μετά ακολουθεί η πολιτική αστάθεια. Ναι, πιο πράσινε μεταφορέ, αλλά δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε αυτό με το να απορρίψουμε την πρόταση τη Κομισιόν. Ευχαριστώ, Φερέιρα. Χαίρομαι που λαμβάνω το λόγο στο τέλος της συζήτησης διότι ήθελα να θίξω δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ε, να πω ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία αποκλειστικά στην ποιότητα των ε, καυσίμων αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας για να ασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό μας σε καύσιμο εντάξει η ποιότητα έχει σημασία αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τον ε, ανεφοδιασμό μας γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική που θα μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των καυσίμων αλλά παράλληλα θα μας διασφαλίσει την, τις εισαγωγές μας, τον εμποδιασμό μας. Μέχρι το 2020 θέλουμε να αυξήσουμε τα κονδύλια που θα χορηγηθούν στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να αυξήσουμε το τμήμα των μελετών που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε την κατάλληλη διοξείδη του άνθρακου. Ευχαριστώ. Ναι, Δεν σα ζήτησα να λάβετε το λόγο, ευαισθητούς βρισκόστε στο κατάλογο ούτω ή άλλω. Επερχόμαστε στον κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ναι, όντω. Ε, έχω το λόγο. Ε, η πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων αποτελεί μια αντίφαση σε σχέση με τη ρητορική της για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την μετάβαση σε μια οικονομία με μικρή κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακου. Θέλουμε να προωθήσουμε τις μη συμβατικές ε, τα μη συμβατικά καύσιμα και υποτιμάμε τις εκπομπές ε, καυσαερίων και αερίων θερμοκηπίου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πόροι εξαντλούνται και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν οι πόροι αυτοί να γίνουν πολύ ε, προσεκτικά θα πρέπει να τύχουν πολύ προσεκτική εκμετάλλευση. Ε, το δεδομένη τη ε, υπογραφή ε, του πρωτοκόλου για την εξάντληση των πόρων, πρώτα στην αλλά και μετά στην Λισαβόνα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για κατάλληλη διαχείριση. Τώρα, σύμφωνα με το Καρδιάη, τον λόγο έχει η κυρία Μόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητάω λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η οδηγία να αλλάξει ριζικά και να αποκλείσει τα oil sands για τις ε, αρνητικότατες επιπτώσεις που έχουν. Μιλάω εξ μια μιας περιοχής ε, της Σαρδινία όπου υπάρχει με ένα δηληστήριο ιδιωτικό που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτήν την ασφαλτούχο την ασφαλτούχο άμμο και αυτό πρέπει να ότι πλήττει σημαντικά το περιβάλλον. Δίνω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Μουέντας. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση και ε, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι με αυτή την ε, πρότασή μας πρόκειται να πετύχουμε ε, του στόχου όσον αφορά τη μείωση του 6% των προβλεπτικών αερίων με το 2020. Ο δε στόχο για να υπάρξει με αυτή την οδηγία μια ποιότητα καυσίμων είναι το να ε, μπορέσουμε να ε, ρυθμίσουμε τι, τι καύσιμο θα έχουμε για τι οδικέ μεταφορέ. Δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε κάποιο συγκεκριμένο καύσιμο. Αλλά αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι το να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται με τα βλαπτικά αέρια του θερμοκηπίου. Οπότε εδώ πέρα έχουν εκφραστεί από όλες τις διαφορετικέ διαφορετικές ε, απόψεις. Ε, μας είπατε για τις εμπορικές ε, συμφωνίες, για τη διαφοροποίηση των αποθεμάτων, το ότι θα πρέπει να ισχύσει η οδηγία και μετά το 2020, οπότε και εγώ όλα αυτά τα οποία είπατε θα τα διαβώσω στον Άρια Σκανιέτα, τον αρμόδιο συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, κύριε Πίτροπε, εμείς σας ευχαριστούμε για τώρα. Έλαβε πέρα η συζήτηση, οπότε πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διατάξης, το οποίο είναι και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων μεταφορών. Floor to the Commission, Commissioner